Συνάδελφοι, αρχίζουμε τις εργασίες μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, Γιάκοπ Ζούμα, τον πρόεδρο της Νοτιού Αφρικής, που παρά τις ε, υποχρεώσεις που είχε στις Βρυξέλλες, τις πολλές υποχρεώσεις, βρίσκεται εδώ μαζί μας. Και μεταξύ άλλων συμμετέχει στις εργασίες μας και η Επιτροπή Ντεβε η αντιπροσωπεία με τις, για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νοτιού Αφρικής και η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος θα πρέπει να φύγει στις 10, 10 5 το αργότερο διότι έχει μία συνάντηση με τον ε, βασιλιά του Βελγίου και γι' αυτό θα πρέπει να περιορίσουμε τις ε, παρεμβάσεις μας. Θεωρούμε ότι οι σχέσεις μας είναι πολύ σημαντικές, όχι μόνο διμερός, αλλά μέσα στα πλαίσια κοινών δεσμεύσεων για τον διάλογο και την ειρήνη στην Αφρικανική Ήπειρο. Και για να αντιμετωπίσουμε τις ε, βασικές προκλήσεις όπως οι κλιματικές αλλαγές. Άρα θα θέλαμε να ε, γνωρίζουμε ποιες είναι οι απόψεις του ως προς τις σχέσεις με την Ευρώπη και ποιο ρόλο θα διαδραματίσει η Νότιος Αφρική μέσα στα πλαίσια των πολύπρευλων διαπραγματεύσεων και των σχέσεων με τα Ηνωμένα Έθνη. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να του δώσω αμέσως το λόγο για να παρεμβεί. Έχετε 10 με 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Ανάπτυξης, Κυρίε και κύριοι πρόεδροι των αντιπροσωπιών με την Νότια Αφρική και τον Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψή μου σε αυτό το κοινοβούλιο, σε αυτό το χώρο και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Μπούζεκ για τη θερμή υποδοχή που μου επεφύλαξε και την, στη διάρκεια της συνάντησης που είχαμε σήμερα το πρωί συζητώντας για θέματα αναπτυξιακής ε, συνεργασίας, τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, τη συνεργασία με την Νότια Αφρική που συνεχίζεται της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εξελιχθεί από την εποχή που ανακτήσαμε ε, τη δημοκρατικό μας καθεστώς πριν από 16 χρόνια. Χθες είχαμε μια σύνοδο κορυφής μεταξύ Νοτιού Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα επιτυχής που έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μια, ένας εταίρος στον τομέα των επενδύσεων και της αναπτυξιακής βοήθειας πολύ σημαντικός για την Νότια Αφρική. Η συνεργασία μας εξελίσσεται πολύ καλώς και καλύπτει τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, το εμπόριο, την επιστήμη και την τεχνολογία Τομεί στου οποίους συνεργαζόμαστε στα πλαίσια συγκεκριμένων έργων και προγραμμάτων. Εκτιμούμε το γεγονός ότι από το 1994 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει δώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για πάνω από 40 έργα τα οποία συμπλήρωσαν τις προσπάθειες της κυβέρνησής μας σε, πιο, σε κρίσιμους τομείς για την ανάπτυξή μας όπως ε, ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, της ενέργειας, ανάπτυξη των υποδομών, υποστήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικροδάνεια. Επενδύσεις σε έργα υποδομής μας επέτρεψαν να φιλοξενήσουμε το παγκόσμιο κύπελο της FIFA Εκτός από τις διμερείς της ε, σχέσεις, ε, η Νότια Αφρική συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της ε, κοινότητας της Νοτιότερης Αφρικής και στην ομάδα των χωρών της Καραϊβικής και της, του Ειρηνικού. Όλες αυτές οι δράσεις και οι σχέσεις επιβεβαιώνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για την, ανάπτυξη, την περαιτέρω ανάπτυξη του αναπτυσσόμενου κόσμου. Η εταιρική σχέση, οι συμπράξεις με την Αφρική και τις άλλες αναπτυσσόμενες περιοχές του πλανήτη πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί ώστε να συμπληρώσει τις αναπτυξιακές προσπάθειες των περιοχών αυτών. Η τρίτη Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει στη Λιβύη θα είναι μια ευκαιρία και για τις δύο πλευρές να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευση και την προσήλωσή τους στην εταιρική σχέση και να δουν πώς μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση ε, σημαντικών στρατηγικών μετά το 2010. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αναξιοποιητές δυνατότητες οι οποίες θα μπορούν να ενισχύσουν την εταιρική μας σχέση με πολύ θετικά αποτελέσματα για την Αφρική. Προσβλέπω σε μία επικοδομητική σχέση η οποία θα μας επιτρέψει με ρεαλιστικό, δημιουργικό τρόπο να δώσουμε νέα όθηση στη σχέση μας, στην εταιρική μας σχέση. Τα αποτελέσματα της ε, διάσκεψης ε, επανεξέτασης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών είναι πολύ σημαντική και για την εφαρμογή της ε, κοινή αναπτυξιακής στρατηγικής πέρα από το 2010. Οι σχέσεις με την Αφρική, τις χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού είναι πάρα πολύ σημαντικές ειδικότερα δε στον τομέα του εμπορίου. Οι δυσκολίες που, αντιμετωπίστηκαν, που αντιμετωπίζονται στην ε, ισχύουσα, στις διαπραγματεύσεις για την ισχύουσα συμφωνία εταιρικής σχέσης έχουν δείξει ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν. Η Σύνοδος Κορυφής που έγινε το 2007 στη Λισαβόνα εξέτασε διαμακρών αυτό το θέμα και όμως δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε πάλι στην ίδια κατάσταση. Ως μέλος της ΣΑΝΤΑΚ και της ομάδας θέλουμε, επιδιώκουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, αλλά πρέπει ωστόσο να επαναλάβω ότι πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες σε μια τελική αναπτυξιακή συμφωνία η οποία θα υποστηρίζει τις προσπάθειες για περιφερειακή ολοκλήρωση και ενοποίηση στην, Νότια Αφρική, στην Νοτιότερη Αφρική, στη Μεσημβρινή Αφρική. Οι κανόνες για, σε ό,τι αφορά την προέλευση πρέπει επίσης να προσδιοριστούν και να επιτευχθεί συμφωνία. Η ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχα θα επιτρέψει στο παγκόσμιο εμπόριο να είναι πιο δίκαιο και να υποστηρίξει το αναπτυξιακό πρόγραμμα άνω των δύο τρίτων των ε, χωρών μελών του ΠΟΕ. Κυρίες και κύριοι, πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να διαδραματίσει κρίσιμο σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση και εποπτεία και παρακολούθηση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο με την Νότια Αφρική, αλλά με το σύνολο της Αφρικής, της Υπήρου και όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη η οποία θα συμβάλλει σε καλύτερη κατανόηση ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσμου και ειδικότερα της Αφρικής. Κατά συνέπεια, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε θέματα εσωτερικά, εσωτερικής, περιφερειακής και παγκόσμιας σημασίας. Προσβλέπουμε στην, ε, ε, στην επίσκεψη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου στη χώρα μας και εκτιμούμε τις πολύ καλές σχέσεις που διατηρούμε με τις αντιπροσωπείες ε, για τις σχέσεις με την Νεότια Αφρική και τον Παναφρικανικό Κοινοβούλιο που καλύπτει και υπάρχει, και, εκτός, και υπάρχει επίσης και η κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση των χωρών των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι Όλοι αυτοί οι οργανισμοί συμβάλλουν σε καλύτερη κατανόηση μεταξύ των χωρών μας. Η παγκόσμια κρίση και η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, κυρίες και κύριες, έχουν δημιουργήσει ανάγκη για την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα από βιώσιμες ουσιαστικές συμπράξεις που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των χωρών μας. Ε, διευρύνουμε ε, και ενισχύουμε την ε, εταιρική μας σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πιστεύουμε ότι η σχέση αυτή μπορεί να παραμείνει ισχυρή και να συμπληρώσει την, τις αναπτυξια... και να στηρίξει τις αναπτυξιακές μας προσπάθειες εφόσον υπάρξει απαιτούμενη δέσμευση και από τις δύο πλευρές προς όφελος τόσο της Νότιας Αφρικής όσο και των λαών της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ για τη θερμία υποδοχή που με απεφυλάξετε και για τον χρόνο που μου διαθέσατε. Αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και δεν έχω έτσι τη δυνατότητα να αναφερθώ σε άλλα σημαντικά θέματα. Θα πω απλώς ότι κατά την άποψή μας η δημοκρατία μπορεί να ε, ενισχυθεί και να κυριαρχήσει εάν οι βουλευτές ως εκπρόσωποι των λαών έχουν τη δυνατότητα να ε, υψώσουν, τη φωνή τους και να φροντίσουν για την πρόοδο των λαών τους. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος σας, γι' αυτό θα πρέπει να είμαι πολύ αυστηρός. Θα ήθελα να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας αυστηρά. Δίνω το λόγο στον κύριο Στρίφλερ, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Την κυρία, ο, καθένας έχει δύο λεπτά παρέμβασης έτσι ώστε να μπορούν να παρέμβουν όλοι. Κύριε Πρόεδρε, η Νότιος Αφρική είναι μία αναπτυσσόμενη χώρα, αλλά είναι μία από τις χώρες BRIC, δηλαδή μία από τις αναδυόμενες χώρες. Πώς βλέπετε το ρόλο σας στην Αφρικανική Ήπειρο και πώς βλέπετε το ρόλο σας ως ε, οθητήρια δύναμη για την ανάπτυξη. Πώς κρίνετε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια ε, δρά στη χώρα σας και πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτής της βοήθειας στα επόμενα έτη. Σας ευχαριστώ. Uh, Ο κύριος Κάσμαν, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τις σχέσεις με την Νότια Αφρική. Ε, ευχαριστώ πολύ. Επειδή ήδη συναντήθηκα με τον πρόεδρο Ζούμα, δεν θα λάβω το χρόνο. Δεν θα λάβω το λόγο. Ο κύριος Γκάλερ, πρόεδρος της Επιτροπής για τη σχέση με το Παναφρικανικό Συμβούλιο. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Oui, Κύριε Πρόεδρε, ξέρουμε ότι διαδραματίσατε σημαντικό ρόλο διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένες σειράξεις στην Αφρικανική Ήπειρο θα ήθελα να τονίσω την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε. Εάν δεν είχατε διαμεσολαβήσει δεν θα είχε εξελιχθεί η κατάσταση όπως εξελίχθηκε παρά το γεγονός ότι παραμένουν πολλές, πολλά σκοτεινά σημεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει περιορισμούς προς τη Ζιμπάμπουε και θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω κατά πόσο αυτό βοήθησε, ήταν καθαρά αντιπαραγωγικό. Σβένσον. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι ε, υπάρχουν σχέδια που αφορούν 60.000 μαθητές που προσπαθούν να καταπολεμήσουν και τον φορέα HIV. Αυτό το είδαμε στην περιφέρεια Ζουλού Νατάλ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πόσο είχε συνεισφέρει η Σουηδία. Ο φορέας HIV και το AIDS είναι μία μάστιγα στην Νότια Αφρική και σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο. Έχετε νέες ρηξικέλευθες ιδέες έτσι ώστε να σταματήσετε την νόσο. Επίσης θα ήθελα να φράσω την, ε, τις ευχαριστίες μου διότι ε, ήδη από την εποχή του Νέλσον Μαντέλα ε, είχαμε προβάλλει βοήθεια από πλευρά Σουηδίας και θέλαμε πάντα να βοηθήσουμε την νοτιοαφρικανική κυβέρνηση. Ελπίζω ε, αυτές οι σχέσεις που έχουμε με την νοτιοαφρικανική κυβέρνηση να επαυξηθούν. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ο ε, Νέλσον ε, Μαντέλα δεν είναι ήρωας μόνο της Νοτιού Αφρικής, αλλά ήρωας της ανθρωπότητας και εν πάση περιπτώσει είναι δικός μου ήρωας. Βεβαίως όλη η ανθρωπότητα στάθηκε στο πλευρό του. Τώρα υπάρχει μία ε, ε, γυναίκα στην Αιθιοπία η οποία θεωρείται ο Μαντέλα της Αιθιοπίας. Μπορεί κάτι να κάνει η Νότιος Αφρική για αυτή την ιδιαίτερα θαραλέα γυναίκα. Κύριος Βότσον, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο Σούμα και να πω πόσο εντυπωσιαστήκαμε πολλοί από εμά από την πρόοδο της χώρας του τα τελευταία χρόνια και του εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του. Ελπίζουμε όλοι η νέα συμφωνία που επετέφθη μεταξύ Νοτιοαφρική και Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε τη σχέση μας και να βελτιώσουμε ε, τη συνεργασία μας, κυρίω σε παγκόσμια θέματα. Ωστόσο, Πρόεδρε Ζούμα, ανησυχούμε λίγο ορισμένοι από εμά από κάποιες εκθέσει που διαβάζουμε για ε, νέα νομοθεσία ενδεχομένως για τον τύπο που φέρεται να περιορίζει την ελευθερία των δημοσιογράφων. Θα μπορούσατε να μας σχολιάσετε αυτές ε, τις φήμες και να μας διαβεβαιώσετε ίσως ότι η ελευθερία του τύπου θα εξακολουθεί να είναι σημαντική στη χώρα σας. Η κυρία Ευχαριστώ. Ε, ως αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας με τη Νότια Αφρική χαίρομαι που παρευρίσκεστε εδώ κύριε Ζούμα και είπατε ότι η δημοκρατία και ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι ζωτικής σημασίας για, το, για τους λαούς. Είχατε μία ζωηρή συζήτηση στη Νότιο Αφρική τον προηγούμενο ε, μήνα σε σχέση με τον ρόλο της πληροφόρησης, της ελεύθερης πληροφόρησης και το ρόλο της δικαιοσύνης. Το ANC συνεδρίασε τον προηγούμενο μήνα το Αφρικανικό Κογκρέσο και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για ε, τις του κυρίου Βαν Ρομποϊ να ε, σταματήσει τις, ε, τις, τους διάφορους περιορισμούς και κυρώσεις που υπάρχουν έναντι της ε, Ζιμπάμπουε. Ο κύριος Βανόρντεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον πρόεδρο Ζούμα με τη σειρά μου. Στο παρελθόν η Νότιος Αφρική δεν προέβαλε ηγετικό ρόλο στο, στη Μεσημβρινή Αφρική. Και εδώ πάλι σκέφτομαι ιδιαίτερα τη Ζιμπάμπουε. Ξέρουμε ότι υπήρξαν εξελίξεις, εξελίξεις τα τελευταία χρόνια και είναι γεγονός ότι η Νότιος Αφρική ε, έχει κάπως ησυχάσει έναντι της ε, ε, Ζιμπάμπουε υπό την ηγεσία του Μουγκάμπε, όπου υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Ξέρουμε ε, πρόσφατα τι γίνεται στα αδαμαντοριχεία του Μαράγκε. Ορισμένοι συνάδελφοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν στόχοθετημένες ε, κυρώσεις. Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι κυρώσεις δεν ε, κατευθύνονται κατά τη Ζιμπάμπουε, αλλά κατά του Γκάμπε και των υποστηρικτών του που έχουν εκμεταλλευτεί τους ε, κατοίκους τα τελευταία δέκα χρόνια. Ελπίζω η Νότιος Αφρική να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για αλλαγές στη ε, Ζιμπάμπου. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Ναι, ευχαριστώ. Ε, και εγώ να καλωσορίσω τον Πρόεδρο. Ήθελα να ρωτήσω κατά τον ίδιο ποια είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα του και θέλω να μας πει κάτι σε σχέση με τις ε, εγκαταστάσεις ε, που δημιουργήθηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ποια δυνατότητα έχει σήμερα το κράτος να τους ε, αξιοποιεί και συνακόλουθα θέλω να μάθω για τους χιλιάδες ανθρώπους που χρησιμοποιήθηκαν είτε σαν φρουροί είτε σε άλλες εργασίες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων όπου ε, τους είχαν υποσχεθεί ένα συγκεκριμένο μισθό αλλά με την λήξη των Ολυμπιακών αυτοί οι άνθρωποι απελήθηκαν και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν πήραν τους μισθούς τους και είναι σήμερα σε απεργίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ως Φλαμανδός ενδιαφέρομαι ανέκαθεν ε, για θέματα Νοτιοαφρικής. Έχουμε και μια συγγένεια γλωσσική, ε, τα Ολλανδικά και τα Αφρικάνς. Και στη Φλάνδρα ε, για την ωραία σας χώρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς και μεγάλη ανησυχία. Και συγκεκριμένα για κάποιο είδος εγκληματικότητας και ιδιαίτερα τις δολοφονίες λευκών ε, αγροτών από το 1994 πάνω από 3.000 δολοφονούνται ε, στα αγροκτήματά τους ε, λευκοί αγρότες με φρικτό τρόπο και δεν είναι τυχαίο, δεν νομίζω. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι διαρθρωτικό το πρόβλημα και υπάρχουν ορισμένες τάσεις που το ε, υποδαβλίζουν. Υπάρχουν οργανώσεις τύπου Kill the Boor, Kill the Farmer, σκοτώστε τον αγρότη ε, και ε, υποκινούνται αυτά τα φαινόμενα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, στο παρελθόν τι κάνατε και τι προτίθεστε να κάνετε στο μέλλον για να εξαφανιστούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Uh, Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ε, θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσα να μας πείτε δύο λόγια για την ειρηνευτική διαδικασία ε, στη Νότια Αφρική και πώς προωθείτε την ειρήνευση σε μια τόσο ταραγμένη ήπειρο σε όλη την Αφρική και στο, στο Βόρεια Αφρική. Ευχαριστώ. Eh, και εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη χώρα όπου μπορούν να επιληθούν πολλά προβλήματα. Υπάρχει όμως ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά την εγκληματικότητα και την ασφάλεια. Και αυτό το θέμα μπορεί να είναι πολύ σημαντική τροχοπέδη για την ανάπτυξη μιας μεγάλης χώρας όπως η Νότιος Αφρική. Θα ήθελα να πω τι σχέδια έχετε εγκρίνει ή θα εγκρίνετε για να αντιμετωπίσετε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η ασφάλεια. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω και εγώ από πλευράς μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θαυμάσιο το Μοντιάλ που διοργανώσατε στη Νότια Αφρική και αποκομίσαμε και πολύ χρήσιμες εμπειρίες και συγχαρητήρια γιατί είδαμε μια άλλη εικόνα για τη Νότια Αφρική και όχι τη συνηθισμένη που βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης. Το οικονομικό όφελος για τη Νότια Αφρική το έχετε υπολογίσει. Γιατί Διαβάζοντας εκθέσει, επιστώνουμε ότι τα λεφτά τα έβγαλαν ε, τα ε, συμφέροντα των πολυεθνικών, η FIFA και τα γήπεδα. Εσείς ε, έχετε αποκομίσει όφελος, το έχετε μετρήσει. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι βρίσκομαι σε ένα κοινοβούλιο με την πληθώρα των ερωτήσεων που μου υποβλήθηκαν, αλλά πολλές από τις ερωτήσεις θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρες να απαντηθούν, αν πρέπει να απαντήσω σε όλους, έτσι ώστε να αποσαφηνίσουμε την κατάσταση. Θα πρέπει να αρχίσω με τη Ζιμπάμπουε, φαντάζομαι γιατί υποβλήθηκαν πολλές ερωτήσεις για τη χώρα αυτή και μετά θα επεκταθώ σε άλλα ζητήματα. Γιατί βλέπω ότι εδώ δίπλα σφυροκοπείται, άρα θα πρέπει να είμαι κι εγώ πολύ προσεκτικός. Για το θέμα της Ζιμπάμπουε θα ήθελα να πω τα εξής. Η Νότιος Αφρική συμμετείχε στη ε, διαδικασία ειρήνευση, ας το πούμε, από τότε που άρχισαν οι ταραχές. Όταν ανέκυψε το πρόβλημα αυτό των ταραχών, η κυβέρνηση Νοτιού Αφρικής παρενέβη. Κάναμε πολλά τότε, τα οποία ε, δεν είχαν αντιληφθεί οι πάντες, διότι δεν θέλαμε να επεκταθεί το πρόβλημα είχαμε συμμετάσχει σε υπουργικές διασκέψεις για να σταματήσει το πρόβλημα. Γιατί ξέραμε ότι θα υπήρχε μεγάλος αντίκτυπος και στην Νότιο Αφρική. Για μας λοιπόν δεν ήταν μόνο ένα ζήτημα να ξέρουμε τι γίνεται στη Ζιμπάμπουε, ήταν ένα θέμα που βρισκόταν πολύ κοντά σε μας. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η Νότιος Αφρική δεν ε, ε, είχε ηγετικό ρόλο. Εμείς κατήχαμε αυτό το ρόλο πριν από οποιονδήποτε άλλον, αλλά ήταν πολύ δύσκολο, διότι οι δύο πλευρές ήταν αποφασισμένες να ε, συνεργαστούν αλλά και να λάβουν υπόψη τις δικές τους πεπιθήσεις. Ο πρώην πρόεδρος, ο Μπέκη, ο κύριος Μπέκη, είχε προσπαθήσει να προβάλλει μία παρέμβαση και προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ρήτρες, συνταγματικές ρήτρες σε σχέση με την καταμέτρηση των ψήφων. Γι' αυτό ε, υπήρξε μεγάλη αυστηρότητα κατά την ε, καταμέτρηση. Αυτή ήταν και η παρέμβαση του πρώην Προέδρου Μπέκη. Και η καταμέτρηση έπρεπε να αρχίσει από τα εκλογικά κέντρα. Γι' αυτό είχαμε σαφέστερα αποτελέσματα. Και πολλές φορές αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι ορατές. η ΣΑΝΤΕΚ προσπάθησε να διευκολύνει αυτή την καταμέτρηση και επήλθε και συμφωνία, συμφωνία την οποία βοήθησε, για την οποία βοήθησε η Νότιος Αφρική. Πολλοί περίμεναν ότι ότι η Νότιος Αφρική θα επικρίνει τη Ζιμπάμπουε, θα εναντιωθεί στη Ζιμπάμπουε. Εμείς αποφασίσαμε να μην το κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να δράσουμε αποτελεσματικά. Γιατί δεν έχει νόημα η κατακραυγή, έχει σημασία η παρέμβαση. Και εμείς πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας αυτή έφερε αυτά αποτελέσματα. και υποβάλαμε μία έκθεση οκτώ εβδομάδες πριν στη ΣΑΝΤΕΚ. Μία έκθεση η οποία κατέδειξε ότι επετελέστη μεγάλη πρόοδο στη Ζιμπάμπουε με έναν οδικό χάρτη και ένα χρονοδιάγραμμα για το τι χρειάζεται να γίνει. Τότε η ΣΑΝΤΕΚ έκρινε τα εξής ότι επειδή θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις, θα πρέπει να κάνουμε έκκληση στην παγκόσμια κοινότητα να άρει τις κυρώσεις έτσι ώστε να δώσουμε μία δυνατότητα σε αυτή τη διαδικασία. Διαδικασία παρέ, παρέμβασης και ειρήνευσης. Βεβαίως ε, πιστεύουμε ότι η κατάσταση δεν είναι η ίδια με αυτήν που ίσχυε στην αρχή ως προς την επιβολή των κυρώσεων, που επέβαλε την επιβολή των κυρώσεων. Εάν αρκεστούμε στις ε, κυρώσεις που εσείς ε, λέτε ότι είναι περιορισμένες. Εμείς θεωρούμε κυρώσεις, όχι περιορισμούς. Τότε το επιχείρημα σε επίπεδο Ζάνο ΠΙΕΦ είναι ότι ενώ η, η κυβέρνηση την χάνει υποστήριξης, ορισμένα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου μπορούν να επιτελέσουν την εργασία τους και μπορούν να ταξιδέψουν ανά τον κόσμο, διότι αυτοί που πλήττονται από τις κυρώσεις δεν μπορούν να ταξιδέψουν, άρα δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν την ενωτική κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που προβάλλεται. Φαίνεται για σας πολύ κάτι το πολύ περιορισμένο, περιορισμένης εμβέλειας. Μην ξεχνάτε όμως ότι οι υπουργοί περιορίζονται και δεν μπορούν να ταξιδέψουν ανά τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα, εάν δεν αρθούν οι κυρώσεις, γιατί περί κυρώσεων πρόκειται, τότε παίζουμε τον, το παιχνίδι εκείνων που θέλουν να παραμείνουν οι εντάσεις στη Ζιμπάμπουε. Άρα θα υπάρχει ολοένα και διονγκούμενη ένταση και οι εκλογές της εκλογές θα υπάρχει βία. Αν αρθούν αυτά τα επιχειρήματα δεν μπορεί κανείς να πει ότι υφίσταται πρόβλημα. και οι κυρώσεις δεν βοηθούν στην εργασία της ΣΑΝΤΕΚ. Αν αρθούν όμως θα υποβοηθηθεί η κατάσταση, διότι η ΣΑΝΤΕΚ δεν μπορεί να δράσει. Εάν δράσει θα σήμαινε ότι συντάσσεται με αυτούς που αντιτάσσονται στην κατάσταση της Ζιμπάμπουε. Άρα έρεται το έργο της ΣΑΝΤΕΚ κατά αυτόν τον τρόπο. Η Νότιος Αφρική έχει 3 εκατομμύρια κατοίκων της Ζιμπάμπουε, υπηκόων μάλλον της Ζιμπάμπουε. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, το γνωρίζουμε. Ξέρουμε και τη δράση Ζάνο ΠΙΕΦ. Ξέρουμε τη δράση της αντιπολίτευσης. Ξέρουμε λοιπόν ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε για να επιλύσουμε τα προβλήματα στη ε, ε, Ζιμπάμπουε. Άρα κάνουμε μια έκκληση στην παγκόσμια κοινότητα να άρει τις κυρώσεις ή να τις αναστείλει τουλάχιστον έτσι ώστε να μην υποσκελίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Στις ε, διαπραγματεύσεις υπάρχει δούνε και λαβίν πιστεύουμε ότι η παγκόσμια κοινότητα θα μπορούσε να δράσει έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Ακόμα και αν δεν πιστεύετε κάτι τέτοιο, αποτελεί τροχοπέδι ε, στη δραστηριότητα της Άντεξ στη Ζιμπάμπουε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η πρόοδος που επιτελείται θα μπορούσε να μην προχωρήσει εξαιτίας αυτών των εμποδίων. Και πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα αδιέξοδο κατά αυτόν τον τρόπο. Και ένας γενικός εισαγγελέα μπορεί να δράσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείτε να θυσιάσετε ολόκληρη τη χώρα. Και θα πρέπει να μας βοηθήσετε να βοηθήσουμε εμεί τη Ζιμπάμπουε στα προβλήματά της. Εμείς έχουμε πληγή από την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην περιφέρεια. Και εμείς προσπαθούμε να διευκολύνουμε την κατάσταση. Χρειάστηκε να επεκταθώ σε αυτό το ζήτημα, διότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους πάντες. Για μας δεν είναι θεωρητικό το ζήτημα, είναι ζωτικής σημασίας και πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε. Ας έρθω τώρα στο θέμα του της προσφυγής ε, του εφετείου για τον τύπο. Το ψήφισμα λέει ας διερευνήσουμε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ένα θεσμός, ένα τέτοιο θεσμικό όργανο. Είπαμε ας διερευνήσουμε, ας διερευνήσουμε το θέμα. Ας διερευνήσουμε το θέμα. Υπάρχει μια τέτοια απόφαση η οποία εμφανίζεται σαν να πρόκειται να θεσπίσουμε ένα νόμο. Θέλουμε τη συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης επειδή ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνει ο τύπος τα μέσα ενημέρωσης προχωράει πιο πέρα από αυτό που θα ανέμενε κανείς πρέπει να σέβονται τα μέσα ενημέρωση την αξιοπρέπεια και την ιδιωτική ζωή των κατοίκων σύμφωνα με το Σύνταγμα. Το κυβερνών κόμμα έχει την ευθύνη, την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των πολιτών γίνονται σεβαστά, προστατεύονται όπως προβλέπει το Σύνταγμα. δεν θέλουμε να καταργήσουμε τους υφιστάμενους θεσμούς. Η τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης παραδέχθηκαν ότι δεν είναι τέλεια και γι' αυτό σκεφτόμαστε να λάβουμε αυτή την απόφαση. Ο Ombudsman, ο συνήγορος του πολίτη, στις περισσότερες περιπτώσεις λέει σε κάποια μέσα ενημέρωση ζητήστε συγγνώμη. Εάν τη συγγνώμη δεν με ικανοποιεί, επειδή εγώ εθίγην, τι να κάνω ως πολίτης της χώρας. Δεν μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματά μου. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής. Πρέπει να υπάρχει ένα δικαστήριο, ένα όργανο στο οποίο να μπορεί κανείς να ασκήσει προσφυγή. Εάν δεν είμαι ικανοποιημένο σαν πολίτης, πρέπει να έχω αυτή τη δυνατότητα. Εξετάζουμε λοιπόν το θέμα και λέμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια διότι δεν μπορεί να γίνεται κατάχρηση της ελευθερίας. Ακόμα όλοι, τα πάντα ρυθμίζονται και ελέγχονται. Γιατί να υπάρχει αυτή η απόλυτη ελευθερία στον, ε, στα μέσα ενημέρωσης που δεν χρησιμοποιείται σωστά, ενώ υπό έλεγχο βρίσκονται ακόμα και οι βουλευτές. Δεν λέμε λοιπόν ότι βαρεθήκαμε πια την ελευθερία του τύπου. Την θέλουμε διότι είναι πάρα πολύ σημαντική για την κοινωνία, αλλά πρέπει να είναι μια ελευθερία που ασκείται σωστά. Σε ό,τι αφορά τα κρατικά μυστικά, υπάρχει νομίζω κάποιο στοιχείο υπερβολής και η συζήτηση που έχει γίνει αφορά το πόσο μπορεί κανείς να προχωρήσει και υπάρχει ήδη ένας νόμος που προστατεύει τις πληροφορίες, τις κρατικές πληροφορίες, διότι υπάρχουν μυστικά, τα οποία, κρατικά, τα οποία πρέπει να προστατεύονται. Αλλά όσοι σχολιάζουν το θέμα έχουν υπερβάλει την κατάσταση. Το νομοσχέδιο έχει ήδη πάρει σάρκα και οστά αλλά το θέμα του δικαστηρίου, όπως είπα, είναι κάτι το οποίο ακόμα βρίσκεται υποσυζήτηση, δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση. Για εκείνους που εργάστηκαν για τις υποδομές, για τα έργα, για το παγκόσμιο κύπελο, υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα για την ανάπτυξη των υποδομών που καλύπτει και αυτή την περιοχή. Και λέμε ότι αυτά τα έργα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και έχουμε προβλέψει και, και τον, τα απαιτούμενα κονδύλια. Θα απορροφηθούν λοιπόν στα προγράμματα, τα έργα αυτά, στα προγράμματα τα οποία πρόκειται να υλοποιήσουμε. Εφόσον ο Πρόεδρος δεν έχει ακόμα χρησιμοποιήσει το σφυρί του... Έχετε όσο χρόνο θέλετε. Α, ναι, θαυμάσια. That's wonderful. Um, the of... Σε ό,τι αφορά ε, το ρόλο που θεωρεί η Νότια Αφρική ότι μπορεί να διαδραματίσει στην Ήπειρο, εμείς πιστεύουμε ότι ε, δεδομένου του μεγέθους, της ανάπτυξης και της εμπειρίας της χώρας έχουμε να διαδραματίσουμε ένα ρόλο πάρα πολύ χρήσιμο, τον οποίο και παίζουμε. Είμαστε σε κάθε ταραγμένο σημείο της Αφρικής και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην ειρήνευση, να σταματήσουμε τη βία. Ε, συμμετέχουμε σε αποστολές ε, διατήρησης της ειρήνης, ε, διαμεσολάβησης και διευκόλυνσης ως χώρα. Χρησιμοποιούμε τεράστιους πόρους προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό το ρόλο θεωρούμε ότι έχουμε. Ότι ε, είμαστε ακριβώς εκείνοι που πρέπει να διευκολύνουμε την Αφρική να ορθοποδήσει σε πολλά θέματα. Ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι ε, είμαστε σε δεύτερη μοίρα γιατί έχουμε και τη δυνατότητα και την ικανότητα και την εμπειρία να βοηθήσουμε σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε ό,τι αφορά τον HIV και το AIDS, βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα και υπήρξαν στο παρελθόν. Κατά τα άλλα, δεν οφείλονταν τα προβλήματα αυτά ε, στις δικές μας πολιτικές. Ήταν πάρα πολύ ορθές οι πολιτικές μας. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι πολιτικοποιήθηκε το AIDS και ο HIV, ο ιός. Δηλαδή, κάποιοι προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τα προβλήματα και τα, και τα μέτρα μας, γιατί είχαν ορισμένοι κάποιες απόψεις που θέλησαν να κυριαρχήσουν στη συζήτηση. Εμείς ε, έχουμε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δραστήριο πολέμησης του HIV και του AIDS και μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Κάναμε δοκιμές δημόσιες, συνεχίζονται αυτές. Ε, τονίζουμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν την κατάστασή τους ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Γιατί μετά είναι απόρριτο το θέμα του καθενός προσωπικό. Αλλά ενθαρρύνουμε όλους να κάνουν τεστ για το AIDS και να γνωρίζουν την προσωπική τους κατάσταση. Και συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα, όπως και πολλά άλλα, άλλωστε, σε σχέση με αυτό. The lady... Σε ό,τι αφορά την κυρία που έχει ε, φυλακιστεί στην Αιθιοπία, βεβαίως δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες. Καλά, καλό είναι να λέμε ότι είναι σαν το Μαντέλα, Εγώ ξέρω το Βαντέλα και όλη του την προσωπική δράση. Δεν γνωρίζω της κυρίας αυτής ε, τη δράση. Μπορεί να έχουμε τις απόψεις μας, αλλά δεν ξέρουμε αν κάποιος άνθρωπος παραβίασε τον νόμο της χώρας του. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε οριστικά σχόλια και κατηγορηματικά. Ε, εφόσον δεν γνωρίζουμε. Αν ήταν ο Μαντέλα, συμφωνώ και προσυπογράφω όλα όσα είπατε. Σε ό,τι αφορά τους Ολυμπιακούς. Και βέβαια προσβλέπουμε σε ε, αυτούς να ε, διοργανώσουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ήδη είχαμε υποβάλει υποψηφιότητα στα μέσα της δεκαετίας του 90 δεν κερδίσαμε. Τώρα είμαστε πολύ ισχυροί και πιστεύουμε ότι θα μας υποστηρίξει αυτή τη φορά η παγκόσμια κοινότητα το αίτημά μας. Θυμήστε μου σε ποια ερώτηση δεν απάντησα. Ε, σας παρακαλώ, διαβάστε μου εδώ τι έχω γράψει. Well, with regard to the economic... Α, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ωφέλη. Ε, του Μουντιάλ του 2010 είναι τεράστια. Τεράστια. Η υποδομή που αναπτύξαμε ε, στην προετοιμασία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου είναι τεράστια. Ε, βελτιώσαμε αεροδρόμια, αυτοκινητοδρόμους. Χτίσαμε γήπεδα. Βελτιώσαμε άλλα στάδια και έπιασαν τόπο τα χρήματα. Ό,τι επενδύσαμε απέδωσε στο ΕΠ μας και χαιρόμαστε. η οικονομική μας ανάπτυξη δεν θα ε, ξανά είναι ποτέ τέτοια όπως φέτος. Αλλά επίσης παρουσίασε την Νότια Αφρική στον κόσμο. Ορισμένοι δεν γνώριζαν καν ότι είχε τις δυνατότητες αυτές η Νότια Αφρική. Το αποδείξαμε. Δείξαμε τις δυνατότητες που έχουμε να ε, τηρούμε χρονοδιαγράμματα, να διοργανώνουμε ε, και μάλιστα μήνες, τέσσερις μήνες έτοιμοι πριν και οι αξιωματούχοι της FIFA ε, που ήρθαν και έκαναν τις επιθεωρήσεις ήταν ικανοποιημένοι. Αλλά έχουμε και την ικανότητα να διοργανώνουμε μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις. Ήταν εκπληκτική αυτή η προσπάθεια. Και τελικά δείξαμε και καταλάβαμε πώς το Μουντιάλ ένωσε την Νότια Αφρική. Επανήλθε το πνεύμα του Μαντέλα της δεκαετίας του 90. Κανείς δεν αμφέβαλε στην Νότια Αφρική. Όλοι ύψωναν τη σημαία της χώρας και όλοι αισθάνονταν πάρα πολύ περήφανοι που είναι Νότια Αφρικανοί. Για μας ήταν τεράστια επιτυχία και οικονομικά και πολιτικά και ε, από πλευρά συμφιλίωσης του λαού. I have not I think uh, we have tried. Let me just. Α, ένα τελευταίο έλεγχο να κάνω. Νομίζω απήντησα. Oh, violence on farm. Α, μάλιστα, η βία κατά των αγροτών. Ναι, όντως αυτό είναι ένα τμήμα της, επικου... της ε, συγγνώμη, εγκληματικότητας ε, στη Νότια Αφρική. Και ξέρετε ότι η εγκληματικότητα είναι κάτι το οποίο καταπολεμούμε και στην Ήπεθρο και στα αγροκτήματα. Έχει συζητηθεί ε, και το συζητούν οι αγρότες με την αστυνομία. Έχει καταρτιστεί ένα σχέδιο με το οποίο είναι ικανοποιημένοι και οι ίδιοι αγρότες. Ε, χρειάστηκε να καταρτιστεί ειδικά για αυτή την περίπτωση. Το έγκλημα έχει κάπως μετριαστεί, έχει κάπως κατευναστεί, έχει γίνει μια μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες η οποία δείχνει ότι ε, καταφέρνουμε να περιορίσουμε το έγκλημα. Είπα για την ειρηνευτική διαδικασία μάλιστα. Άλλη ερώτηση που δεν απέντησα. Παρακαλώ θυμίστε εκείνη που κάνατε ερωτήσεις γιατί... Ε, όχι, απαντήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, α εγκρίνουμε τη μερίσια διάταξη. Επανερχόμαστε στο σημείο 1 ε, μετά ε, την απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Δεν θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τον Παύλο Κλίμκιν, υφυπουργό εξωτερικών υποθέσεων και τον Μπόρις Ταραζούκ, πρόεδρο της Επιτροπής για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας. Από τις 17 θα συζητηθούν αυτά τα θέματα. Το διευρυμένο Προεδρείο, το οποίο προβλεπόταν για το απόγευμα, θα, γίνει, θα συνεδριάσει σήμερα στις 11 και 4. Εγκρίνουμε και τα πρακτικά ε, των συνεδριάσεων της Δευτέρας Σεπτεμβρίου 6ης και 7ης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά. Δεν υπάρχει αντίρρηση, άρα εγκρίνονται. Punto successivo, conclusione διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Τουρκμενιστάν. Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Η πρόταση ψηφίσματος για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Τουρκμενιστάν. Ε, έχει ως εισηγήτρια αυτή η πρόταση ψηφίσματος την Όρικα Νικολάη και βασιζόμαστε σε δύο διαφορετικά έγγραφα. Το ε, έγγραφο σύστασης της ε, θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το επίμαχο ζήτημα και το δεύτερο μία πρόταση ψηφίσματος που συνοδεύει τη σύσταση για να εξετάσουμε την πρόταση σύσταση, γνωμοδότησης για να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς τη Σύμφωνη Εταιρική Σχέση αυτή. Δίνω το λόγο στην κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα. Ώστε αυτά τα οποία θα πω να είναι απόλυτα σαφή. Σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος θέλησα να εξασφαλίζει η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που χρειάζεται το Τουρκμενιστάν που είναι η δημοκρατική υποστήριξη και αυτά που χρειάζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να υποστηρίξει στην ευρύτερη γειτονία της δημοκρατική και οικονομική σταθερότητα που είναι κάτι του αναγκαίο και για τις δύο πλευρές. Πρόσφατα η ανάπτυξη του Τουρκμενιστάν οφείλεται ε, και στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της χώρας σε έτσι ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τους πολίτες της. Μετά από τις επισκέψεις μου στο Τουρκμενιστάν είχα την ευκαιρία να συζητήσω όχι μόνο με ε, ε, υπεύθυνου της κυβέρνησης αλλά και με πολίτες με το διπλωματικ... με το εκπροσώπους του διπλωματικού σώματος επίσης. Και θα ήθελα να σας πω ότι σύμφωνα με τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει η Ευρώπη πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία με τη ε, χώρα αυτή, η Κεντρική Ασία πρέπει να συμπεριληφθεί στα προγράμματα συνεργασίας μας διότι αυτό είναι προς όφελος των οικονομικών μας συμφερόντων αλλά και μία δυνατότητα για μας να εξασφαλίσουμε την αναγκαία δημοκρατική σταθερότητα ώστε να υπάρξει ασφάλεια στην ευρύτερη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν κάθε συμφέρον να υπογραφεί, να συναυθεί αυτή η συμφωνία, διότι δεν μπορούμε να εμπλακούμε ως ενεργοί εταίροι με άλλο τρόπο, αν δεν υπάρχει δηλαδή το απαραίτητο νομικό πλαίσιο. Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουρκμενιστάν πρέπει να στηρίζεται στο κατάλληλο ε, νομικό πλαίσιο, στην κατάλληλη νομική βάση που θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα αυτού του διαλόγου και αυτής της συνεργασίας. Υπάρχουν ε, ορισμένες προκαταλήψεις που ε, αφορούν τον τρόπο ενημέρωσης. Το Τουρκμενιστάν δεν ε, αποτέλεσε ούτε αποτελεί αυτό που αποτελεί Νότια, Νότια Κορέα σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το Τουρκμενιστάν με τα υψηλά δημοκρατικά, τις υψηλές δημοκρατικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά οι πρόοδοι που έχουν γίνει μετά την αλλαγή του, του καθεστώτος πρέπει να τονιστούν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εκείνοι που παίζουν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τον εκδημοκρατισμό της χώρας προέρχονται από τις δομές του ΟΗΕ το ΟΗΕ είναι παρόν στη χώρα μέσα από διάφορα προγράμματα όπως, το πρόγραμμα, όπως και τα προγράμματα του Europa House και πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε και να συμβάλλουμε στην ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών στη χώρα αυτή και στις προσπάθειες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν και στην ευρύτερη περιοχή. Χαιρετίζω την παρουσία των ΜΚΟ η οποία συμβάλλει στην ε, εφαρμογή των υψηλών αρχών για την ε, διατήρηση του διαλόγου. Είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω, να συνεργαστεί με όλους τους σημαντικούς γείτονές της και το Τουρκμενιστάν είναι ένας σημαντικός γείτονας της κεντρικής, στην Κεντρική Ασία. Οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλα σημαντικά πολιτικά συμφέροντα στην ε, περιοχή όπως η Ρωσία που έχει παράδοση συνεργασίας οικονομικής και άλλης με την ε, περιοχή, όπως και η Κίνα, το Τουρκμενιστάν είναι ανοιχτό όμω σε μια ευρύτερη συνεργασία με όλες αυτές τις χώρες και στον ΟΗΕ ο πρόεδρος, ε, ε, στο βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος υπογράμμισε την επιθυμία της χώρας του να συνεργαστεί με όλες τις χώρες και για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε τη σύναψη αυτής της συμφωνίας επιτρέποντας το Τουρκμενιστάν να παίξει σημαντικό ρόλο στην Κεντρική Ασία, μια περιοχή και που πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα μαζί με το Τουρκμενιστάν της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την έναρξη ισχύω τη ε, ε, συνθήκη τη Λισαβόνα και τη δημιουργία τη υπηρεσία εξωτερική δράση θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η παρουσία, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Νικολάη. Έχουμε αρκετούς εγγεγραμμένους και αρχίζουμε από τους Κιώδης. Πέτερλε από το ΕΛΚ. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εργασία της εισηγήτριας. Νομίζω ότι τα κατάφερε πολύ καλά και ήταν πολύ υπεύθυνη η προσέγγιση της. Κατανοώ βεβαίως το δίλημά της και τις τελικές της υποδείξεις έτσι ώστε να ορίσουμε μία νομική βάση συνεργασίας με αυτή την χώρα της Κεντρικής Ασίας. Γιατί με αυτή τη χώρα δεν υπάρχει βάση συνεργασίας, νομική βάση. Ασχοληθήκαμε με θέματα προτεραιότητας, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και νομίζω ότι αυτή η έκθεση περιλαμβάνει ό,τι πρέπει να περιληφθεί και τονίζουμε την τήρηση των αξιών και αρχών που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο μιας παρόμοιας συμφωνίας. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία του συνέρχεστε, ελευθεροτυπία και ούτω καθεξής, καθώς και ένα κράτος δικαίου. Οι μη κυβερνητικέ όμως δεν μπορούν να δράσουν σε αυτή τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αντιπροσωπεία στη χώρα αυτή και ακόμα και ο Ερυθρός Σταυρός δεν μπορεί να λειτουργήσει στο Τουρκμενιστάν από όσο γνωρίζουμε. Οι γιατροί χωρίς σύνορα εγκαταλείπουν επίσης το Τουρκμενιστάν. Υπάρχουν προβλήματα για να ταξιδέψουν οι κάτοικοι στην Λοδαπή και οι μη κυβερνητικέ αντιμετωπίζουν ένα πολύ δύσκολο έργο, δεν μπορούν καν να δράσουν. Άρα, είτε θα περιμένουμε έτσι ώστε να συναυθεί αυτή η συμφωνία και να συμβεί κάτι το θετικό σε αυτή τη χώρα, μετά από τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια, ίσως ε, κάτι γίνει ή η άλλη επιλογή είναι να συνεχίσουμε με τη σύναψη έτσι κι αλλιώς. Θα πρέπει να επέλθει μια συμφωνία, να συναυθεί η συμφωνία και γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την, αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές ε, γιατί τουλάχιστον θα υπάρχει νομική βάση για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας καλύτερα από ό,τι μπορούμε μέχρι τώρα. Προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι κάθε ε, χώρα στην ε, Κεντρική Ασία θα πρέπει να θεωρηθεί ως ε, περιφέρεια ύψης της στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να αναλάβουμε μεμονωμένα μικρά ε, βήματα για να βελτιωθούν τα πράγματα. Άρα υπ' αυτή την έννοια ε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη για να μπορέσουμε να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία κύριος Μπέλντερ από την ομάδα του. Την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε σήμερα ε, το θέμα του Τουρκμενιστάν, αλλά δεν είναι καινούριο. Εδώ και χρόνια ε, εκρεμεί. Και καταλαβαίνω αυτά που λέει και η συγχύτρια. Δεν είναι εύκολο να μάθουμε έγκυρες πληροφορίες ε, και στην Ανατολική Ευρώπη δεν γνωρίζουμε πολλά για το Τουρκμενιστάν. Διάβασα ε, με πολύ ενδιαφέρον την έκθεση και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Και υπάρχει ένας δισταγμός εδώ. Ε, αλλά αν συσφίξουμε τις σχέσεις μας με το Τουρκμενιστάν, αυτό θα είναι ε, υπέρ ε, της βελτίωσης κατάστασης του πληθυσμού. Αλλά ε, τι γίνεται με την ελευθερία της έκφρασης, την ανεξιθρησκεία και την ελεύθερη λατρεία. Και δυστυχώς από την εποχή του Νιασόφ, του ε, Τουρκμενμπάξι μέχρι σήμερα δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα και αυτό το λένε πολλές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και επί τόπου. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση για την ε, ανεξιθρησκεία και αυτό δεν ισχύει μόνο για χριστιανούς αλλά και για άλλες θρησκείες. Στην παράγραφο 13 λοιπόν θα είχα να ασκήσω αυτή την κριτική για την έκθεση ήτριας. Με προβληματίζει. Υπάρχει αυστηρός έλεγχος κοινωνικός που δεν το επιτρέπει. Και Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τη σύναψη των σχέσεων ή τη σύσφυξη των σχέσεων μας με το Τουρκμαϊστάν δεν ξέρω κατά πόσο είναι σκόπιμο. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα δίλημα τώρα. Έχουμε κριτική, έχουμε κάποια προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά θα ήταν καλύτερο να έχουμε σχέσεις, να ε, ε, συνάψουμε μια τέτοια συμφωνία και έτσι να βοηθήσουμε για να βελτιωθούν και τα υπόλοιπα που μας ενοχλούν. Ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε την ευκαιρία να διαβολευθούμε και να ε, καταλήξουμε σε κάτι λογικό. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θα ήθελα λοιπόν να βάλω και εγώ αυτή την απόχρωση εδώ για το θέμα της ελευθερίας της άσκησης λατρείας και της ε, είναι απογοητευτικά τα πράγματα και βλέπουμε μια συνέχεια με το παλιό καθεστώς. Δεν έχει διακοπεί αυτή η προβληματική κατάσταση. Ευχαριστώ. La Κυρία Χάουταλα, που είναι πρόεδρος υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Είμαι και σκιώδης εξ ονόματος των Πρασίνων. Νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία για εμάς να αποσαφηνίσουμε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητες που έχει ως προς μια επίσημη σύναψη συμφωνίας, δηλαδή ε, κατά πώς θα συμφωνήσουμε με αυτή τη σύναψη και θα ήθελα να είμαστε σίγουροι για το κατά πόσο θα προωθήσουμε αυτή την Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, δηλαδή κατά πόσο θα δημιουργήσει τους όρους για να ε, προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο εκδημοκρατισμός και το κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα. Και κανένα συνάδελφος ε, μέχρι τούδε δεν αρνήθηκε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε αυτή τη χώρα. Άρα η πρότασή μου είναι η εξής. Εάν συμφωνείτε, θα μπορούσα να προτείνω στους συναδέλφους στην υποεπιτροπή να οργανώσουμε μία ad hoc ακρόαση με την Επιτροπή στις 14 Οκτωβρίου το αργότερο και με ε, ορισμένες εμπλεκόμενες οργανώσεις και βεβαίως θα πρέπει να το εγκρίνει και η συγγήτρια αυτό και η Επιτροπή για να δούμε κατά πόσο μία τέτοια πολιτική θα βοηθούσε στον εκδημοκρατισμό. Άρα θα μπορούσαμε να αναβάλουμε την προθεσμία υποβολής τροπολογιών έτσι ώστε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα και να δούμε πώς έχει η κατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, δηλαδή γύρω στις 16 Οκτωβρίου. Τώρα, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι υπάρχει κάποια σύγχυση σε σχέση με τη νομική βάση για το ε, πώς να αντιμετωπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τουρκμενιστάν. Η νέα ενδιάμεση συμφωνία ετέθη σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2010 και περιλαμβάνει την δυνατότητα συνεργασίας στον τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν λοιπόν έχουμε κάτι περισσότερο από την παλαιά συμφωνία που υπήρχε επί Σοβιετικής Ένωσης από το 1979, αυτό θα ήταν πολύ καλό. Επίσης χρειάζεται η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης πριν ε, συσταθεί, αποσταλεί μία αντιπροσωπεία στο Άσκαμπατ. Ξέρουμε ότι είχε εξευρεθεί μία λύση με άλλες χώρες που βρίσκονται σε παρεμφερή κατάσταση με την αποστολή μιας αντιπροσωπείας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα του στον, τον Απρίλιο του 2009 έθισε πέντε ορόσημα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ενδιάμεση συμφωνία εμπορίου, η οποία έχει τεθεί ε, μόλις σε ισχύ. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα ορόσημα Καταρχήν και αυτό αναφέρθηκε από τον κύριο Πέτερλε. Το Κοινοβούλιο ζήτησε με τη θέση ισχύ αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας εμπορίου όχι το περαιτέρω βήμα, αλλά αυτό Καταρχήν, να επιτραπεί ο Ερυθρός Σταυρό να λειτουργήσει ελεύθερα στο Τουρκμενιστάν, να απελευθερωθούν όλοι οι αντιρρησίε συνήθιση και οι πολιτικοί κρατούμενοι, επίσης να μπορούν να ταξιδεύουν στην Αλοδαπή οι κάτοικοι. Τέταρτον, ελεύθερη κυκλοφορία στι μη κυβερνητικέ και επίσης οι ανθρωπιστικές οργανώσει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο Τουρκμενιστάν ε, προχωρούμε με σοβαρότητα ή μιλάμε για ευσεβείς πόθους και θεωρείτε ότι ένα περαιτέρω βήμα θα επιτρέψει να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα που ήδη ε, ενυπάρχουν στο Τουρκμενιστάν. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά βήματα που έχουν γίνει. Δηλαδή, το Τουρκμενιστάν έχει κυρώσει τις ε, περισσότερες συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, αλλά δεν είμαστε πεπισμένοι ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Και Επίση, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από όσο γνωρίζω, επισκέφθηκε το Τουρκμενιστάν ένα μήνα πριν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει το, τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δεδομένα. Εφόσον λοιπόν είναι παρούσα η Επιτροπή, και θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις μας, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο μπορεί να μας δώσει ε, μία εκτενή ανάλυση για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί έτσι ώστε να πληρωθούν αυτά τα πέντε ορόσημα που ορίστηκαν τον Απρίλιο του 2009 και πώς έχουν ενταχθεί στην ε, συμφωνία ε, εμπορίου και συνεργασίας. Υπάρχει νομική βάση για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση αυτή τη νέα ενδιάμεση εμπορική συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, αλλά θεωρώ εξ ονόματος υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι έπρεπε να θίξω αυτά τα ζητήματα πριν ε, συνενέσουμε στο περαιτέρω βήμα που προτείνεται. Σας ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας και πολύ σοβαρές και αντιρρήσεις. Κλείνει ο κατάλογος των σκιωδών με την συνάδελφο Λόζιν. Ευχαριστώ. Συμφωνώ πολύ σε μεγάλο βαθμό με τις προαλήσαντες, ιδιαίτερα με την κυρία Χάουταλα. Ε, θέλω να την υποστηρίξω ως προς τη διαδικαστική της ε, πρόταση. Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η κυρία Νικολάη τώρα θεωρεί ότι έχει οριμάσει ο χρόνος για να υπογραφεί η συμφωνία. Και εγώ προσεκτικά προσπάθησα να αναλύσω την κατάσταση στο Τουρμενιστάν. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα αλλά έχω πάρα πολλέ αναφορές από μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ανησυχούν βαθύτατα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν. Έστω ότι υπογράφουμε τώρα τη συμφωνία, υπάρχει για μένα κίνδυνος πραγματικός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πέσουν στο βωμό ε, των οικονομικών και γεωστρατηγικών συμφερόντων των κρατών μελών. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή σήμερα δεν θέλω να πω πολλά λόγια, τα είπαν τα περισσότερα. Η δική μας πολιτική ομάδα της ΓΚΟΕ απορρίπτει τη σύναψη συμφωνίας και τονίζω ότι συμφωνώ με τα διαδικαστικά που πρότεινε η κυρία Χάουταλα. Κλείνουν ε, οι παρεμβάσει των σκιωδών. Η κυρία Γκόμας έχει το λόγο. Και μετά στην κυρία Άξελ Νάισα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Γκόμες, καταρχήν. Και εγώ υποστηρίζω κύριε Πρόεδρε αυτά που είπε η κυρία Οπτάλα, η Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι οι πληροφορίες που έχουμε πάρει από τις, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε πάρει από διάφορες πλευρές και η έκθεση η ίδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, δείχνει ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτό το προηγούμενο, διότι θα αποτελέσει πολύ σημαντικό προηγούμενο. Το να ξεχάσουμε για, οικονομικούς λόγους τα ανθρώπινα, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τίποτε δεν εμποδίζει την, την, μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξει στο Τουρκμενιστάν χωρίς μια συμφωνία. Η συμφωνία αυτή θα στήριζε, θα στήριζε πολιτικά ένα καθεστώς το οποίο συμπεριφέρεται σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα με απαράδεκτο τρόπο, δεν επιτρέπει την ελεύθερη λειτουργία πολιτικών κομμάτων, δεν επιτρέπει την ελευθερία του τύπου, δεν επιτρέπει ε, τη θρησκευτική ελευθερία, δεν επιτρέπει στους πολίτες να ταξιδεύουν έξω από τη χώρα, να περιορίζει τις ε, οργανώσεις, τη λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κλπ. Με βάση όλα αυτά, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε ποτέ να δεχθεί σε αυτή τη φάση μια τέτοια συμφωνία. Θα δεχόμουν να πάω στο, στην ακρόαση που πρότεινε και ο Τάλα. Τίποτε δεν εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν ε, ε, σχέσεις με το Τουρκμενιστάν λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μια τέτοια χώρα με τέτοιο ε, ε, ε, που συμπεριφέρεται έτσι σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο εταίρο. Βεβαίω θέλω και εγώ να ακούσω τι έχει να μας πει η Επιτροπή για την επίσκεψή της μετά το Σεπτέμβριο σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 2 της συνθήκης δικαιούται να ενημερωθεί από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ξέρω πώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα να ξέρω εάν ε, γίνονται προσπάθειες να υποστηριχθούν εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς την παρέμβαση των αρχών και τι δραστηριότητες έχει ε, εφαρμόσει στο, ε, Τουρκμενιστάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς για να εξασφαλίσει την προστασία, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν αφορά μόνο το Τουρκμενιστάν. Ε, έχει, αφορά επίσης το μήνυμα που θα μεταφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άλλες συμφωνίες, για άλλες συμφωνίες που βρίσκονται υπό επεξεργασία. με χώρες στις οποίες δεν ισχύει το κράτος δικαίου. Και δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο μία έκθεση η οποία περιέχει στην παράγραφο 7 τη φράση ε, «Λυπάται την... Ε, για τις...» ε, για την ασυνέπεια που έχει επιδείξει το Κοινοβούλιο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι το πιο συνεπές θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχθώ αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση στις, ε, της παραγράφου 7. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να βγω από το ρόλο μου ως ε, Προέδρου καταρχήν και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τις παρεμβάσεις Λέζινγκ Χάουταλα Γκόμες. Τώρα, ως πρόεδρος, δίνω το λόγο στην κυρία Άξελ Νάιζε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Hello. Uh, my name is... Αξέλ λέγομαι. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. από τις αρχές Σεπτεμβρίου εργάζομαι στο γραφείο για το Τουρκμενιστάν. Κατανοώ τις ανησυχίες που εκφράζουν τα μέλη του Κοινοβουλίου που έλαβαν το λόγο για να πούν ότι όντως η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πόρο απέχει από να φτάνει σε οποιαδήποτε ε, διεθνή πρότυπα. Έχουμε απόλυτη επίγνωση του γεγονότος αυτού και δεν προσπαθούμε να κρύψουμε ούτε τις δυσκολίες, ούτε ε, τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι πολίτες του Τουρκμενιστάν. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι κανένα νομικό πλαίσιο μάλλον η έλλειψη νομικού πλαισίου οποιαδήποτε συνεργασία ε, μας εμποδίζει να δράσουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά την άποψή μας χρειάζεται αυτή η συμφωνία πλαίσιο ως εργαλείο για να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Από τεχνικής πλευράς ακόμα επικρατεί η νομική βάση της συμφωνίας του 89 με την τότε Σοβιετική Ένωση. Μια ενδιάμεση προσωρινή συμφωνία που πολύ σωστά τόνισε η κυρία Χάουταλα ε, που τέθησε ισχύ την 1η Αυγούστου φέτος έχει και ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, το θέμα είναι ότι αυτή η ρήτρα δεν είναι νομική βάση για να πούμε σε πολύ συγκεκριμένο διάλογο ούτε ως ε, εργαλείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το Τουρκμενιστάν είναι ένας τρόπος να επαναλάβουμε ότι ε, η ενδιάμεση συμφωνία βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της δημοκρατίας. Αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι νομικά δεσμευτικό, δεν είναι νομική βάση για να προωθήσουμε ένα πρόγραμμα. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε επικοδομητικοί και να προωθούμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, χρειαζόμαστε ένα νομικό εργαλείο στα χέρια μας. Γι' αυτό και η συμφωνία. Και επειδή είναι περιορισμένη η σχέση μας μέχρι τώρα και υπάρχει και απομόνωση και από δική μας πλευράς που συνεχίζεται χρόνια ολόκληρα. Και δεν βοήθησε για να βελτιωθεί πολύ η κατάσταση στο Τουρκμενιστάν, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε. Το 2007 με την εκλογή του νέου Προέδρου Μπέντι ε, Μοχάμετ έγιναν πολλές υποσχέσεις και όπως γνωρίζουμε οι υποσχέσεις αυτές δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο. Ε, μπορεί βεβαίω να υπάρχει μια βελτίωση, μπορώ να σας αναφέρω μερικούς τομείς αν, επιθυμείτε. Έχουμε δει συγκεκριμένη βελτίωση σε ό,τι αφορά ε, τους εσωτερικούς περιορισμούς ε, μετακινήσεων και ταξίδιων στο εσωτερικό της χώρας, παρόλο που δεν έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Υπάρχει ένα ίδρυμα για τη δημοκρατία και το, τα ανθρώπινα δικαιώματα που ιδρύθηκε στο Ασκαμπάτ και έχουμε και με πολλές σχέσεις μαζί τους. Ε, στη συνέχεια ε, συστήθηκε μια κυβερνητική, κρατική καλύτερα επιτροπή ε, για να προσφεύγουν οι πολίτες ό,τι αφορά τη δράση των οργάνων επιβολής της τάξης και το Μάιο του 2010 είχε και μεγάλη μεταρρύθμιση στο νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος εγκρίθηκε και μειώνει τις ε, μέγιστες πηγές, ποινές, συγγνώμη, και ε, αλλάζει και τις κυρώσεις ε, για παραβάσεις του αστικού δικαίου και προχωρεί σε πρόστιμα αντί για προσωποκράτηση. Επίσης, το πολυκομματικό σύστημα και ένα νέο κόμμα έχει εμφανιστεί, το Αγροτικό Κόμμα και επίσης έχουν γίνει ανακοινώσεις και για άλλες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες παρακολουθούμε πολύ στενά και για τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και για τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις και για τη μεταρρύθμιση του τύπου. Ε, λίγα μόνο παραδείγματα κάποιων θετικών ε, ενδείξεων και μεταρρυθμίσεων που βλέπουμε. Βεβαίως δεν ανταποκρίνονται στις δικέ μας προσδοκίες, αλλά βήματα γίνονται. Ε, στις περιορισμένες λοιπόν σχέσεις που έχουμε με τους Τουρκμένους φαίνεται ότι εκείνοι επιθυμούν πραγματικά να ανοίξουν περισσότερο ε, χώρα και να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά το πρώτο που αναφέρουν ως ε, μέλημά τους δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι προφανές αυτό, αλλά πραγματικά θέλουν μια νέα εποχή και έχουμε και θετικά μηνύματα και για το άνοιγμα της χώρας. Επαναλαμβάνω, αν δεν γίνει λοιπόν αυτό το άνοιγμα, θα χάσουμε και εμείς ευκαιρίες να συνεργαζόμαστε με έναν πρωταγωνιστή στην περιοχή. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία βεβαίως δεν τα θυσιάζουμε στο βωμό των οικονομικών συμφερόντων, δεν είναι μόνο οικονομικά τα συμφέροντα, θέλουμε να βοηθήσουμε και τους πολίτες της χώρας αυτής. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να παίξει η χώρα ρόλο στη σταθεροποίηση ε, της περιοχής του Αφγανιστάν και στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Είναι σημαντικό στοιχείο και αυτό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ένα άλλο σημαντικό και δεν σας το κρύβω ότι μας απασχολεί πάρα πολύ είναι η διαφοροποίηση ε, ε, στην προμήθεια ενέργειας για μας. Η μεγάλη πρόκληση είναι να έχουμε ένα ισοζύγιο ειλικρινές και τίμιο μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πρόθεσης των ε, συμφερόντων του λαού, του Τουρκμενιστάν αλλά και των δικών μας ενεργειακών συμφερόντων στην περιφέρεια. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία εκεί. και αν γίνει η συμφωνία αυτή ε, ανοίγει και το δρόμο για το θέμα αυτό. Να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα της κυρίας Χάουτα αλλά τώρα και της κυρίας Γκόμες. Ως προς την πρόσφατη επίσκεψη που αναφέρθηκε στην Ασκαμπάτ τον Ιούνιο έγινε ένας διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συζητήθηκαν και ακαθόδη θέματα για τα ορόσημα που μας είπατε. Ήταν σαφέστατο στο μυαλό μας αυτό. Να έχει πρόσβαση η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού ε, στις φυλακές κρατουμένους με ε, ονόματα κρατουμένων που ε, κατηγορούν ότι υφίστανται βασανιστήρια ε, και κάποια άλλα θέματα άνοιξη θρησκείας ε, συζητούμε με τους Τουρκμένους. Μπορεί να μην είναι εύκολος ο διάλογος πάντα, αλλά υπάρχει, υφίσταται και ήταν ο τρίτος γύρος διαλόγου που είχαμε για αυτό το θέμα. Και όπως είπε η κυρία Γκόμες, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως υπενθυμίστηκε το Τουρκμενιστάν, έχει κυρώσει ε, τις περισσότερες από τις διεθνείς συμβάσεις για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα είναι πώς θα τα εφαρμόσει. Στις περιορισμένες δυνατότητες που έχουμε, στον επόμενο διάλογο ε, που έχει προγραμματιστεί το 2011 στο 2013 έχουν αποφασιστεί ορισμένε δράσεις, μεταξύ αυτών υποστήριξη ε, στο Κοινοβούλιο, στη νομική μεταρρυθμίση, στη Γαλλία Χρηστή Διακυβέρνηση και επίσης ε, θα συνεχίσουμε τις μαζικές προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση στην παιδεία που πιστεύουμε ότι θα προσφέρει και προστιθέμενη αξία και τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Και αν πιστέψουμε τον πρόεδρο, το έχει και στι προτεραιότητες τους. Ελπίζω να μην με ακρηγόρησα, είμαι στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ. Μπορώ να απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις. Ε, πριν τη πριν δώσω το λόγο για τα συμπεράσματα στην εισηγήτρια, στην κυρία Νικολάη, αν συμφωνείτε όλοι, ας αναβάλουμε την προθεσμία υποβολής τροπολογιών, κάτι το οποίο θα αποφασίσει η γραμματεία. Δεν υπάρχει αντίρρηση, άρα έτσι συμφωνούμε. Άρα δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Νικολάη. Uh, Ευχαριστώ. Σε σχέση με την αναβολή υποβολής ε, προθεσμίας, εάν ε, συμφωνείτε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ληφθεί μία απόφαση τώρα, πριν γνωρίζουμε όλα τα, τα στοιχεία. Βεβαίως μιλήσαμε για τα ορόσημα, τα οποία είναι έξι, δεν είναι πέντε, είναι έξι και εν μέρη βρίσκονται στην οδό εφαρμογή στο Τουρκμενιστάν, όμως είναι πολύ μεγάλη ε, η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς και το ε, παρόν. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε μία χώρα. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να επικρίνουμε την έλλειψη δημοκρατικών κριτηρίων. Μπορούμε άρα να απομακρυνθούμε και να επικρίνουμε ή να εμπλακούμε και να υποστηρίξουμε τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Νομίζω ότι το να συμμετάσχουμε στη διαδικασία σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτές τις προδιαγραφές κατά ευφυή τρόπο και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει μία ε, κοινή αντιμετώπιση αυτών των αρχών. Διαφορετικά θα είμαστε ε, δεν θα είμαστε τίποτα άλλο παρά παρατηρητές για να δούμε ότι δεν εφαρμόζονται οι δικές μας αξίες και οι δημοκρατικές προδιαγραφές. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης προ ε, προσχέδιο σύστασης, ε, μάλλον ε, συμφωνίας εταιρική σχέσης συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μολδαβίας. Υπάρχει το σχέδιο σύστασης για τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μολδαβίας. Μιλάμε για τις γενικές αρχές συμμετοχής της Δημοκρατίας της ε, Μολδαβίας, τα προγράμματα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, στο Κισινάου θα γίνει η υπογραφή της ε, συμφωνίας του πρωτοκόλου δηλαδή και εμείς θα πρέπει να αποφανθούμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βότσον για να μας πει πώς έχει το σχέδιο σύσταση. Έχετε το λόγο κύριο Βότσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Πρόεδρε, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μολδαβία διαφέρουν από εκείνε που αντιμετωπίζει το Τουρκμενιστάν, το οποίο μόλι συζητήσαμε και που μας παρουσίασε η συνάδελφος Νίκολάη, αλλά αξίζει και αυτή την προσοχή μας. Η χώρα αντιμετωπίζει τις τρίτες εκλογές της στη διάρκεια δύο ετών μετά, αφού δεν μπόρεσε δύο φορές να επιλέξει πρόεδρο το κοινοβούλιο. Ο κύριος Γκίμπου διέλυσε το κοινοβούλιο και κήρυξε γενικές εκλογές για τις 28 Νοεμβρίου. Μας καλούμαστε να εγκρίνουμε και να λάβουμε θέση για το πρωτόκολλο τη συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μολδαβίας. Οι σχέσεις είναι καλές, θέλουμε να τις ενισχύσουμε, δεν πρέπει να φυστούμε προσπαθειών για να βοηθήσουμε τη Μολδαβία ε, να δείξει ότι μπορεί να προσεγγίσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό να ωφελήσει ε, τους πάντες σε ό,τι αφορά την οικονομική υποστήριξη, την ε, διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων και τις ευρύτερες θετικές επιπτώσεις της συμφωνίας σύνδεσης. Το σχέδιο σύσταση ε, συμβαδίζει με την προσέγγιση, με την προσέγγιση που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζεται στην εταιρική σχέση για τη συμμετοχή σε κοινοτικές υπηρεσίες και κοινοτικά προγράμματα. Η εταιρική σχέση για κάθε πρόγραμμα προϋποθέτει την υπογραφή ενός μνημονίου συναντήληψης που υπογράφεται ανάμεσα στις δύο πλευρές και απαιτεί και μία δέσμευση από τη χώρα που συμμετέχει στην εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει οικονομικά στην στα προγράμματα. Αν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο με τη Μολδαβία όπως ελπίζουμε, χρειάζεται σταθερότητα πολιτική και δημοκρατική πορεία της χώρας για την εφαρμογή του πρωτοκόλου. Η τρέχουσα κατάσταση στη Μολδαβία είναι κάτι που μας απασχολεί αυτό το αδιέξοδο, η Επιτροπή αποφάσισε στο εγγύς μέλλον να στείλει μια ε, αντιπροσωπή ad hoc στη Μολδαβία η οποία θα συναντήσει ανθρώπους ε, από όλες ε, τις πλευρές και θα ενημερώσει κατόπιν την Επιτροπή μας. Νομίζω όμως ότι θα ήταν σκόπιμο να εγκρίνουμε την απόφαση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλου για, την ε, εταιρική για, τη, για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Ευχαριστώ κύριε Βότσον. Μας ε, πείσατε, ήσασταν απόλυτα πιστικός, υπάρχει ομοφωνία ως προς την έκθεσή σας, γι' αυτό κλείνουμε ε, το θέμα τώρα και θα βρεθούμε στις 11 και 4 για το διευρυμένο Προεδρείο. Σας ευχαριστώ. Ritiro quanto detto, relatore Watson. <laughs> Η κυρία Μάκοβεϊ θέλει να παρέμβει. Με συγχωρείτε. Άρα δεν ήμουν και τόσο πιστικός. Ας ακούσουμε τι θα πει η κυρία Μακοβέη. Ελπίζω να μας πείσατε παρόλα αυτά. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να πω για να υποστηρίξω αυτά που είπε ο Γκραμ και άλλη μια φορά να τονίσω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε και τις δημοκρατικές δυνάμεις στις επικείμενες εκλογές ανεξάρτητα από την πολιτική ομάδα στην οποία ανήκουν διότι οι δημοκρατικές δυνάμεις στη Μολδαβία ε, είναι κατά του κομμουνιστικού κόμματος, του κομμουνιστικού και όχι του σοσιαλιστικού κόμματος. Προσβλέπουμε λοιπόν στην επίσκεψή μας εκεί τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Υποστήριζω θερμότατα τις προσπάθειες του συναδέλφου Γότσον ε, και για το γεγονός ότι από τη δική μου χώρα αναλαμβάνονται προσπάθειες για να βοηθηθεί η πολιτική και η κοινωνία στη Μολδαβία. σε μια χώρα που είναι πάρα πολύ φτωχή και στην ίδια μου την πόλη το Σάββατο ε, έγινε μια μεγάλη εκδήλωση και διαδήλωση για τη Μολδαβία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζεται ε, για να βοηθήσουμε τους πολίτες στη χώρα αυτή και θα πρέπει να είμαστε στο πλευρό των πολιτών οι οποίοι ε, ακριβώς ε, δεσμεύονται να βοηθήσουν τον κόσμο σε αυτή τη ε, μεριά της Ευρώπης. Ξέρω κατά πόσο κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ομοφωνία κύριε Βότσον.